Σουδάν θα χρησιμεύσουν για την επόμενη έκθεση, γιατί και εγώ είχα πάει στο Νότιο Σουδάν και τα μαθήματα που θα αντλήσουμε από εκεί θα τα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ωραία, η συζήτηση ολοκληρώνεται και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Ora l'ordine del giorno reca Τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε τη δήλωση ε, της Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία για την κατάσταση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και το λόγο έχει η κυρία Άστον. Ε, thank you very much, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σα είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψει με του Ευρωβουλευτές για τη διαμάχη στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Όταν μαζί με τους Προέδρους ε, Μπαρόζο και Βαν Ρόμποϊ συναντήθηκα με τον Πρόεδρο Μετβέτεφ στην ε, διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας, ο Πρόεδρος Μετβέτεφ ήταν αισιόδοξο ό,τι αφορά την πιθανότητα επιτυχίας της ε, συνεδρίας του Καζάν. Είπαμε στον κύριο Μετβέτεφ ότι υποστηρίζουμε τις προσωπικές προσπάθειες διαμεσολάβησης αλλά και το έργο της ομάδας του Μίνσκ. Οι δηλώσεις της Ντοβίλ των Πρόεδρων Ομπάμα Μετβέντεφ και Σαρκοζή αποσαφήνισαν ότι είναι και η ώρα για επίτευξη συμφωνίας, γιατί διαφορετικά θα τίθεται ένα αμφιβόλο η δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών για ανέβρεση λύσης. Δυστυχώς, παρά τα σημαντικά μηνύματα σε υψηλότερο επίπεδο, η αναμενόμενη επιτυχία της συνεδρίασης του Καζάν δεν πραγματοποιήθηκε. Οι πρόεδροι του Αζερβαϊτζάν και τη Αρμενία δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να καταλήξουν συμβαστική λύση. Οι σχέσει μεταξύ των δύο χωρών είναι δύσκολε. Πρόσφατα, μάλιστα, συνάντησα του υπουργού εξωτερικών και τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν και δεν έχω καμία ψευδέστηση για την περιπλοκότητα αυτών των διαπραγματεύσεων. Οι συμπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, με ενημέρωσαν για, τη δυσκολία, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο έργο τους. Την περασμένη Παρασκευή ενημερώθηκα και από τον ε, Υπουργό Εξωτερικών της ε, Λουθουανίας, που είναι τώρα ο πρόεδρος της ΟΑΣΕ θα πρέπει να βρούμε συμφωνία με βάση τις βασικές αρχές και χαίρομαι που και οι δύο ενδιαφερομένες πλευρές τάχθηκαν υπέρ της διπλωματικής διαδικασίας για την ανέβρεση ειρηνικής λύσης. Θα πρέπει όμως να έχουμε περαιτέρω πρόοδο τους επόμενους μήνες, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για να βρεθεί συμφωνία πριν τα τέλη του έτους και να συμβεί αυτό πριν τις ε, χώριες προτεραιότητες που θα έχουμε το 2012 τι βουλευτικέ εκλογέ στην Αρμενία και το 2013 στο Αζερβαϊτζάν. Η συνέχιση του στάτου κουβό είναι απαράδεκτη. Επίση, απαράδεκτη είναι οποιαδήποτε προσπάθεια να επιληθεί η σύγκρουση ή να επηρεαστούν οι διαπραγματεύσει με τη χρήση βία ή έστω και τη απειλή χρήση βία. Μια ειρηνική διαθέτηση τη διένεξη του Ναγκόνο Καραπάχα εξυπηρετεί και τα στρατηγικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μεταμορφώσει ολόκληρη την περιοχή του Νοτιού Καυκάσου θα χαράξει το δρόμο για μια σταθερότητα πολιτική και περιφερειακή, αλλά και θα δημιουργήσει νέε οικονομικέ ευκαιρίε. Τα σύνορα θα ανοίξουν όχι μόνο μεταξύ Αρμενία και Αζερβαϊτζάν, αλλά και μεταξύ Αρμενία και Τουρκία. Οι δρόμοι, σιδηρόδρομοι και αγωγοί φυσικού αερίου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συντομότερο δρόμο και να συνδέσουν τι χώρε τη περιοχή ακόμη περισσότερο. Ο Νότιο Κάφκασο μπορεί να γίνει αυτό που θα έπρεπε να είναι ήδη μία πύλη μεταξύ τη Ασία και τη Ευρώπη. Όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, σίγουρα είναι και προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και προσυλλομένοι να, ενισχύσουμε, να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες και τις προσπάθειες των συμπροέδρων της ομάδας του Μίνσκ. Οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται από το 1994 με την παρούσα μορφή συνεχίζονται και είναι δυνατή μια συμφωνία. Βέβαια, το είδο τη ε, στήριξη που θα παράσχουμε θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευση με του συμπροέδρους τη Ομάδα Μίνσκ και τι ενδιαφέρομενε πλευρέ και περιμένουμε ε, τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πάντως, ό,τι και αν συμβεί στις τελικές διαπραγματεύσεις ε, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για μας και θα, διαδραματίσουμε, θα διαδραματίσει ρόλο στον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών μας ε, ως προς τις χώρες αυτές. Ο Μύρος Αφλάιτσεκ, ο διευθυντής μας, με εκπροσώπησε σε αποστολή στις χώρες αυτές τον περασμένο μήνα και διατράνωσε αυτό το μήνυμα. Ε, επίσης έχουμε τη, στη Βαρσοβία το Σεπτέμβριο την Σύνοδο Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Εκεί θα δούμε τις δυνατότητες που έχει μια διευρυμένη ε, συνεργασία. Θα πρέπει επίση ε, να υποστηρίξουμε τις, την κοινωνία των πολιτών, τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και να στηρίξουμε αυτέ τι διαπροσωπικές επαφέ ε, και στα πλαίσια του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Αλλά θα μπορούσαμε να εντείνουμε τι προσπάθειές μα. Επίση, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε ιδιαίτερε ευθύνε στην εφαρμογή του διακανονισμού από τη στιγμή που θα φτάσουμε στο στάδιο αυτό σε στενή συνεργασία με του διεθνεί μα εταίρους. Πολλά θα έχουμε να κάνουμε. Ανασυγκρότηση, άρση ναρκοπαιδείων, πρόσφυγες, επιστροφές εσωτερικά εκτοπιστέντων και την πρόθεση της οικονομικής ανάκαμψης και της ασφάλειας. Αναγνωρίζω επίσης και το ρόλο των άλλων εταίρων μας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περιοχή και θα είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με τους περιφερειακούς μας εταίρους ε, όπως την Τουρκία. Πρότεινα το διορισμό νέου ειδικού εκπροσώπου για τον Νότιο Κάφκασο για να να προωθήσει όλες αυτές τις εργασίες σε στενή συνεργασία με τους συμπροέδρους της ομάδας του Μίνσκ. Ίσως το πιο, η πιο σημαντική συνεισφορά μας θα είναι η συνέχιση και η ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων και με την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Η νέα ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία που συζητήθηκε νωρίτερα εδώ προβλέπει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιού Καυκάσου. Νέες συμφωνίες σύνδεσης, Ευρύτερε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ενίσχυση και διευρυμένη κινητικότητα, διατομιακή συνεργασία και συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα και αυξημένη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και της ανοιχτής κοινωνίας. Κυρία Πρόεδρε, ο γενικός μας στόχος είναι να βοηθήσουμε τις γειτονικές μας χώρες να εφαρμόσουν αυτή την πλήρη ατζέντα και θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε και τη διμερή μας συνεργασία προκειμένου να βοηθήσουμε την επίτευξη διακανονισμού. Ο Στέφαν Φίλε πρόσφατα επισκέφθηκε την Αρμενία για να διερευνήσει τρόπους προώθησης των σχέσεων αυτών. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ε, σημαντικό να έχουμε πιο ελκυστικά προγράμματα, πιο στέρεα προγράμματα για να ξεπεράσουμε τις ε, δύσκο, τα δύσκολα κληροδοτήματα του παρελθόντο. Επίση, αυτή είναι η επιλογή που θα πρέπει να κάνουν οι ηγέτε τη Αρμενία και του Αζερβαϊτζάν προ το συμφέρον των λαών του. Γνωρίζουμε ποια είναι η επιλογή που θα θέλαμε να πραγματοποιήσουν. Είναι η επιλογή του συμβιβασμού και τη ε, ειρήνη. και πιστεύουμε ότι μπορούμε να παίξουμε ρόλο υποστηρίζοντας του συμπρόεδρου τη ε, ομάδα του Μίνσκ για να πραγματοποιήσουν αυτή τη φιλοδοξία. Ευχαριστώ κυρία Στον. Εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν εκ μέρους του ΑΛ για δύο λεπτά ο κύριος Μπροκ. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ στο κόμμα του ΕΛΚ, στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, γιατί ανησυχούμε ότι θα υπάρξει νέος ε, ανταγωνισμός, νέα κούρσα εξοπλισμών, στην οποία θα συμμετέχουν δύο όμορες χώρες ε, και αυτό αναγκαστικά θα οδηγήσει σε εμπόλεμη σε σύραξη. Ε, πρέπει λοιπόν να σπάσουμε αυτό τον ε, φαύλο κύκλο για να μην έχουμε αυτό που ζήσαμε πριν από τρία χρόνια στην περιοχή εκείνη όπου ξαφνικά ξέσπασε πόλεμος και δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτούς τους ε, κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας είναι απόλυτα σαφές ε, ότι εμείς ζητάμε την ε, επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους. Και επίσης πιστεύουμε οι έξι αρχές τις οποίες αναφέρει η ομάδα Μίνσκ ε, και που έγιναν αποδεκτές και από τις δύο πλευρές ε, επιτέλους να εφαρμοστούν, να αναζητηθούν άλλα αίτια του γιατί δεν εφαρμόζονται αυτές οι αρχές. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο και ε, δεν ξέρω κατά πόσον ο τρίτος που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι ο ουδέτερος διαπραγματευτής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη πολιτική και όπως έχω ήδη πει και κατά το παρελθόν πρέπει στις χώρες αυτές επιτέλους να προσφέρουμε κίνητρα για πολυμερή προσέγγιση πρέπει να τους πούμε ότι αν συνεργαστούν αυτό θα τους ανοίξει το δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο θα βελτιώσει τις ε, διμερείς τους σχέσεις. Ε, η ιδέα της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν ανέκαθεν να συνδυάζει τα συμφέροντα και με τον τρόπο αυτό να αντιπαρέρχεται την ένταση του παρελθόντος. Νομίζω λοιπόν ότι ε, το θέμα της πολιτικής γειτονίας το έχω αναφέρει στην υπατή ε, εκπρόσωπο. Πάντως όλοι μας ενδιαφερόμαστε η περιοχή αυτή να μην αποσταθεροποιηθεί γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων κάτι το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον μας και για λόγους ασφάλειας αλλά και ανεργειακής πολιτικής. Εκ μέρους των και Δημοκρατών για δύο λεπτά ο λόγος του κ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Άστον, χαίρομαι που συζητούμε το θέμα του Ναγκόρο Καραμπάχ. Πολλοί από εμά ανησυχούν εξαιτία τη ένταση που επικρατεί και κλιμακώνεται. Δεν θέλουμε να ξαναβρεθούμε στην, ε, στην κατάσταση του να φτάσουμε πάλι καθυστερημένοι. Η αποτυχία της Συνόδου του Καζάν μας δείχνει μάλλον ότι η ομάδα του Μίνσκ έχει φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων της. Όμως η βασική ευθύνη για την ε, πύληση της ε, διαφοράς αυτής ε, βαρύνει τους ηγέτες των δύο κρατών. Οι ηγέτες των δύο αυτών χωρών θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα γραφτούν τα ονόματά τους στην ιστορία ως ε, ε, άνθρωποι ε, πώς θα γραφτούν τα ονόματά τους στην ιστορία ως αυτοί που έφεραν δεινά στους πολίτες τους ή αυτοί που έφεραν την ειρήνη. Η δική μας πολιτική γειτονίας αναφέρεται σε αυτή την σε αυτή την σε αυτή τη σύγκρουση ενυπνώση που υπάρχει και το σημαντικό δεν είναι να υποστηρίξουμε τις σχέσεις μας με αυτές τις δύο χώρες, αλλά και τις σχέσεις αυτών των χωρών μεταξύ τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης να παίξει ένα ρόλο για να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Οι εκπρόσωποι αυτών των χωρών έχουν συμμετάσχει δραστήρια, ενεργά, στην ε, συνέλευση της ε, Ανατολής, μαζί με δικούς μας ε, βουλευτές. Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε κοινά φόρα και αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την συνεργασία ανάμεσα στους δύο λαούς. Βασίζομαι και εμπιστεύομαι την Πολωνική Προεδρία, καθώς επίσης και τη Συνοκορφή της ε, Βαρσοβίας, ε, προκειμένου να δοθεί μια καινούργια όθηση ε, στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Ευχαριστούμε κύριε Βικένιν. Εκ μέρου των φιλελευθέρων για 1,5 λεπτό ο λόγος στην κυρία Όγιουλαντ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί εκπρόσωπε, έχουμε πολλά ανησυχητικά μηνύματα από την περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ ε, τον τελευταίο καιρό παρά την εκεχηρία ε, ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν. Ε, θα ήθελα να καλέσω και το Μπακού και το Γερεβάν να μην εμπλέκονται σε εμπόλεμες πράξεις. Στις 24 ε, Ιουνίου είχαμε τη συνάντηση κορυφή στο Καζάν, αποτυχία δυστυχώς, και αυτό είναι μία απόδειξη ότι οι προσπάθειες ομάδας Μίνσκ δεν αρκούν και πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, διότι το Αζερβαϊτζάν και η Αρμενία είναι ε, χώρε που εντάσσονται στην πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επίλυση του προβλήματος. Κυρία Άστον, θέλω να σα ενθαρρύνω να αντιμετωπίσετε την κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη την εδαφική ακαιρεότητα του Αζερβαϊτζάν κυρίως ε, και ιδίως ε, ε, λόγω των τεσσάρων ψηφισμάτων που έχουν εκδοθεί από τα Ηνωμένα επί του θέματος. Είναι προς όφελος ε, και των δύο κρατών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να επιληθεί το πρόβλημα αλλά βέβαια σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο και αυτό θα επιτρέψει να, επανέλθει, να επέλθει η δημοκρατία στο Νότιο Κάφκασο. Ο λόγος για ένα λεπτό στην κυρία Λούναντσεκ εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Άστον, οι παγωμένες συγκρούσεις ε, αποτελούν εμπόδιο ε, στις, ε, στην εταιρική, στις εταιρικές μας σχέσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν που είναι μέλη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Είναι πως καλό την Αρμενία να ξεκινήσει αμέσως την απόσυρσή της από τα κατεχόμενα εδάφη και ταυτόχρονα ζητώ από το Αζερβαϊτζάν να περιορίσει τον ε, αμυντικό του προπολογισμού που είναι υψηλότερο από όλο τον προπολογισμό τη ε, Αρμενία, Οπότε αυτό αποτελεί ε, κίνδυνο να ξεσπάσει ξανά εμπόλεμη σύγκρουση, σύραξη. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια. Τι εσεί τι πιστεύετε, κυρία Άστον. Εγώ προσωπικά πιστεύω θα ήταν πολύ καλό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντικαταστήσει την Γαλλία στην Προεδρία τη ομάδα του Μίνσκ. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο τη θα πρέπει να αντιπροσωπεύεται στην ομάδα του Μίνσκ, όχι μόνο ένα κράτο μέλο. Επίση πιστεύω ότι η αξιοπιστία <clears throat> και η συνέπεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η λογική συνέπεια, <clears throat> τίθεται ένα αμφιβόλο. Να δούμε την Αμπχαζία, την Νότιο Σετία κλπ. Ε, μιλούμε εκεί, ε, μιλούμε για την ε, ε, δαφική ακαιρεότητα, αλλά στον Αγκόνο Καραγάχ μιλούμε για δαφική ακαιρεότητα και ε, αυτοδιάθεση. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας, 1,5 λεπτό για 1,5 λεπτό λόγο στον κύριο Προβέρα. Το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν είναι ευρέως ε, γνωστό ε, γιατί κυρίως υπάρχουν ε, μεροληπτικές ε, πληροφορίες. Όμως ένα πράγμα αδιαμφισβήτητο είναι η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ενός κυρίαρχο κράτους. Επίσης πρέπει να γίνεται σεβαστό το απαραβίαστο των συνόρων, η περίπτωση Γεωργίας, Μολδαβίας, Κύπρου και κατόπιν τούτου και Αζερβαϊτζάν την σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπήρξαν πολλέ ε, τοποθετήσει. Έχουμε τη δήλωση του Ελσίνκη του 2008, ε, τη δήλωση του ε, Συμβουλίου Ασφαλείας και το Κοινοβουλίο μα έχει τοποθετηθεί επί του θέματο. Η εδαφική κυριότητα ενό κυρίαρχου κράτου διασφαλίζεται από το διεθνέ δίκαιο και το να αμφισβητείται αυτή η αρχή, αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνει κανεί μεροντικέ εμπόλεμε συγκρούσει αποτέλεσμα την αποστεθεροποίηση ολόκληρου του κόσμου. Η Ευρώπη έχει ιδιαίτερα συμφέροντα και ενδιαφέρον για τον Αγκόνο Καραμπάχ, διότι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν μπαίνουν στην πολιτική γειτονία όπου προβλέπεται η σταθερότητα και η συνεργασία ανάμεσα σε χώρε εταίρου. Άρα δηλαδή πρέπει να εργαστούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να σα υπενθυμίσω ότι η θέση τη Αρμενία, η κατοχή επί των εδαφών, σκαφών του Αζερβαϊτζάν με τον χρόνο παγιώνεται και αυτό δυσχεραίνει το να, ε, να αναζητηθεί και να επιτευχθεί λύση στην περιοχή. Για τους μία εγγεγραμμένους για 1,5 λεπτό λόγο στον κύριο Στογιάνοφ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω με τους δύο προηγούμενους ομιλητές γιατί η αιτία της σύγκρουσης ε, αποτελεί ε, ε, ε, η αιτία της σύγκρουσης ήταν η απόφαση των Μπολσεβίκων του, στη δεκαετία του 20 του προηγούμενου, του, του, προηγούμενου αιώνα να αποσπάσουν ένα κομμάτι από την Αρμενία και να το παραχωρήσουν στο Αζερβαϊτζάν. Το ίδιο έγινε και με, την, με το μακεδονικό έθνος. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα μέχρι και σήμερα. και η Βουλγαρία και η Ελλάδα χάρη στην ε, συνεπή τους ε, θέση απέφυγαν να ε, δημιουργηθούν παρόμοια προβλήματα με την αυτοποκαλούμε δημοκρατία της Μακεδονίας και στα Βαλκάνια, αλλιώς θα είχαμε τα ίδια προβλήματα και εκεί. Ε, κυρία Άστον, εσείς λέτε ότι οι σιδηρόδρομοι και η πετρελαγωγή θα πρέπει να περνά, να, να κάνουν τη μικρότερη δυνατή διαδρομή, αλλά οι γείτονε τη Αρμενία την αποκλείουν. Ε, θα πρέπει να το καταγγείλουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Στογιάννοφ. Παίρνουμε στου λοιπού ομιλητέ. Για δύο λεπτά ο κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλό το ότι αυτή τη συζήτηση για τον Αγκόρνο Καραμπάχ την κάνουμε πριν από το καλοκαίρι και κατά την άποψή μου θα ήταν καλύτερα ως Κοινοβούλιο να είχαμε θεσπίσει ψήφισμα και να στείλουμε χειρό μήνυμα προς όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οφείλω να ομολογήσω ότι ανησυχώ ε, για το ότι σε αυτή την περιοχή επικρατεί ένταση. Ε, υπάρχει κίνδυνος ε, ένας από τους δύο να χάσει την ψυχραιμία του και ο άλλος ή ο ίδιος να επωφεληθεί ε, γεωστρατηγικά. Βεβαίως εμείς δεν πρέπει ε, να ε, πάρουμε το μέρος της μίας της άλλης πλευράς. Οφείλουμε να καλέσουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους σε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Επειδή λοιπόν το καθεστώς δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει, υπάρχει κίνδυνο σε μία από τις δύο πλευρές να εγκαταλείψει σωστό δρόμο. Η Ρωσία είναι ο προμηθευτής ε, και των δύο κρατών ενδεχομένως υπάρχει μια κρυφή ημερήσια διάταξη όπου αν υπάρξει σύγκρουση αυτός θα εμφανιστεί ως ειρνοποιός αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο ανησυχώ διότι εμείς ε, στην περιοχή ε, μπορούμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα από άλλους εμπιστοσύνη, προστασία των μειονοτήτων δημιουργία δημοκρατικών θεσμών οικονομικός εξυγχρονισμός συμπερίληψη σε κοινό οικονομικό χώρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ε, αν εμπλακεί θα προσφέρει τα μάλα και στις δύο πλευρές ε, και χαίρομαι κυρία είπατε εκπρόσωπε που το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλήσατε και με τις δύο πλευρές διότι το Καζάν απέτυχε διότι η Ρωσία ίσως να μην είναι τίμιος διαπραγματευτής γι' αυτό λοιπόν αυτό το κενό δεν πρέπει να το αφήσουμε ε, ακάλυπτο και πρέπει να αναζητήσουμε την προοπτική της ε, συμφιλίωσης. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Κυρίλο. Ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε με συντριπτική πλειοψηφία το ψήφισμά του για την ανάγκη νέα ε, ευρωπαϊκή στρατηγική για την Νότιο Κάφκασο. Στο ψήφισμα υπογραμμίζουμε τη στρατηγική σημασία αυτή τη γειτονική περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κίνδυνο από τι παγωμένε συγκρούσει όπω του Ναγκόνο Καραμπάχ. Και κίνδυνο υπάρχει όχι μόνο για τα εμπλεκόμενα τμήματα, αλλά για την ευρύτερη περιοχή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πληθυσμό που ε, επηρεάζεται από, το, από τη σύγκρουση αυτή, εξακολουθεί να ζει στο φόβο και περίπου ένα εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισθέντων είναι όμοιροι αυτής της κατάστασης ε, και χρειάζεται ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Όντως, η ομάδα του Μίνσκ και προσωπικά ο πρόεδρος Μετβέντεφ ε, έκαναν πολλές προσπάθειες για ειρηνευτική επίλυση. Γιατί όμως ε, προσκρούμε σε διέξοδο κάθε φορά που οι εμπλεκόμενες πλευρές κάθονται στη τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Επίσης, ε, ο απόρριτος χαρακτήρας των διαπραγματεύσεων νομίζω ότι έχει φτάσει στα όρια του. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν αποφασίσουν οι χώρε να συμφωνήσουν και αν ξεσπάσει πόλεμο, δεν μπορούμε να μείνουμε αμέτωχοι παρατηρητέ. Επίση, θα πρέπει και η Γαλλία με τον εκπρόσωπο της στην ομάδα του Μίσκ να ασκήσει πιο δραστήριο ρόλο μαζί με τη Ρωσία και τη ΣΥΠΑ να ασκήσει ε, πιέσει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν με τις βασικές αρχές. Επίσης θα πρέπει να δοθούν ε, χέγγια ασφάλειας και στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές όπως ζητήθηκε για να εξασφαλιστεί ε, και να εδραιωθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει κίνητρα σε ό,τι αφορά τις υποδομές, την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις ώστε ο κόσμος στην περιοχή ε, και οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπιστέντες να γυρίσουν τις αιστείες τους και να δουν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα της ειρήνης. Πριν από ένα χρόνο υποστηρίξαμε ένα ψήφισμα για μια ασφαλέστερη γειτονία. Κάτι τέτοιο θα εξασφαλίσει μια μόχλευση ώστε να δημιουργήσουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια των ενεργειακών αγωγών στην Ευρώπη. Κυρία Στον, κυρία είπατε εκπρόσωπε, πρέπει επιτέλους να πάτε και εσείς προσωπικά στην περιοχή και να εμπλακείτε ενεργά στην στην απεμπλοκή αυτών των παγωμένων συγκρούσεων που γίνονται όλο και πιο θερμές. Κύριε Κυρίλοφ, ο κύριος α, σήκωσε μπλε κάρτα. Δέχεστε την ερώτηση. Ναι, λέει ο κύριος Κυρίλοφ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο κύριος Κυρίλοφ γνωρίζει ότι η Ρωσία είναι αυτή που προμηθεύει κατεξοχήν όπλα στην εμπόλεμη αυτή περιοχή έχει και βάσεις, πολύ, πολλά, πουλάει όπλα και νομίζω ότι αυτή ήταν η μεγάλη επένδυση του Πρωθυπουργού <laughs> Πούτιν στην ειρήνη της ε, νοτιού, του Νοτιού Καυκάσου και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ναγκόνο Καραμπάχ. Το γνωρίζετε αυτό κύριε Κυρίλοφ. Ευχαριστώ. Όντως είναι δύσκολη ερώτηση που θέσατε το ομολογώ, αλλά το ενδιαφέρον στην περίπτωση αυτή είναι ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη Ρωσία να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι είναι και μακροπρόθεσμα προς το συμφέρον της Ρωσίας να διευθετηθεί αυτή η σύγκρουση. Παρόλο που ορισμένες δυνάμεις στη Ρωσία θεωρούν ότι βραχυπρόθεσμα συμφέρει τη Ρωσία να κρατήσει και τις δύο χώρες, Αζερβαϊτζάν και Αρμενία, στη σύγκρουση αυτή. Εγώ πιστεύω ότι είναι δυνατή η επίλυση της σύγκρουση. Αλλά χρειάζεται φυσικά και ενεργό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη στρατηγική εταιρική σχέση που έχουμε με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο Σεγγέντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φέτος στις 11 Απριλίου είχαμε μια πρωτοβουλία προκειμένου το Ουγγρικό Κοινοβούλιο να καταδικάσει την αρμενική επίθεση στον Αγκόνο Καραμπάχ το 1992 και η Ουγγαρία να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου να θέσει ως προτεραιότητά της την επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Το Αζερβαϊτζάν έχασε 20% της επικράτειάς του και χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένα εκατομμύριο χρειάστηκε να, να, να γίνουν πρόσφυγες. Η γενοκτονία ε, στον Αγκόνο Καραμπάχο ε, ήταν κάτι αντίστοιχο με την αρμενική ε, γενοκτονία. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ορισμένες γενοκτονίες και να θυμάμαστε άλλους και να χρησιμοποιούμε διπλά μέτρα και σταθμά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να επιληθεί ειρηνικά το πρόβλημα και η σύγκρουση στον Αγκόνο Καραμπάχ. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό το λόγο κύριο Κοβατσέφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Άστον. Η σημερινή συζήτηση προκλήθηκε από την αυξανόμενη ένταση και τις τριβές καθώς και τα θύματα που έχουμε καθημερινά στον Αγκόνο Καραμπάχ. Θα πρέπει να εκτονωθεί αυτή η ένταση και να σταματήσουμε αυτές τις επιθετικές φρασεολογίες. Είναι παράδεκτο οι ηγέτες της περιοχής να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους απαγωμένες συγκρούσεις για να ενισχύσουν την ομοιοποίησή τους. Θα πρέπει να βρούμε μια ειρηνική λύση στη σύγκρουση του Ναγκόνο Καραμπάχ με σεβασμό της εδαφική εκκαιρεότητας και με μη χρήση βία. Αυτέ οι αρχέ είναι πολύ βασικέ στο διεθνέ δίκαιο. Και εγώ ανησυχώ για αυτή την κούρσα εξοπλισμών που γίνεται και την αγορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Κάτι τέτοιο απειλεί την ειρηνική διευθέτηση τη σύγκρουση αυτή και αφήνει ανοιχτέ τι πόρτε για τη χρήση βία. Κάτι που δεν θα εξυπηρετήσει κανένα σε τελική ανάλυση. Η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να καταλήξουν σε συμβαστικέ λύσει και να σταματήσουν εμένα πεισματικά στα στο δική του ε, θέση. γιατί θα βγουν και οι δύο χαμένοι τελικά από μια έλλειψη από μια έλλειψη συμφωνίας και ειρηνευτικής επίλυσης. Και οι περιφερειακές δυνάμεις θα πρέπει να διαδραματίσουν το ρόλο τους ε, στις διαπραγματεύσεις και να ενισχύσουν τις επαφές τους με τις χώρες αυτές. Και η Ρωσία και η Τουρκία θα πρέπει να δείξουν οριμότητα και να ξεπεράσουν τις μακεβελικές ε, αρχές και διαχωρισμούς για να καταλήξουμε σε ειρηνική διευθέτηση. Τέλος, περιμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη διπλωματική της παρουσία και ρόλο και χαίρομαι για το διορισμό του νέου ειδικού απεσταλμένου στο Νότιο Κάφκασο γιατί χρειαζόμαστε μια ειδική πολιτική, ιδιαίτερη πολιτική για κάθε χώρα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της. Δεν βλέπω την κυρία Χέρτσοκ στην αίθουσα, οπότε δίνω το λόγο για 1,5 λεπτό ο κύριος Τόκες. Mr. Τόκες, Mr. Τόκες. Έχετε το λόγο κύριε Τόκες. Τόκες. I'm sorry um, Κύριε Τόκε, λυπάμαι που διαταράζω αυτή τη ρομαντική σκηνή και στιγμή, αλλά πρέπει να σας δώσω το λόγο. You can resume afterwards, but... Μπορείτε να συνεχίσετε μετά προς το παρόν. Πάρτε το λόγο παρακαλώ. floor, Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη. Μην ανησυχείτε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Συνάδελφοι, πριν από τη Σύνοδο Κορυφή του Καζάν του Ιουνίου, του 24 Ιουνίου, η διεθνή ε, κοινότητα είχε εκφράσει πολλέ ελπίδε για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν επί του προβλήματος του Ναγκόνο Καραμπάχ. Μια περιοχή στην οποία κατοικούν εδώ και αιώνες χριστιανοί Αρμένοι και τουρκικής προέλευσης μουσουλμάνοι Αζέρι. Ε, Πλάι-πλάι ζούσαν στο νότιο Κάφκασο για πολλά, πολλούς αιώνες υπό διάφορα καθεστώτα. Δυστυχώς δεν επετέφθη η συμφωνία. Ε, αντίθετα χάθηκαν όλες οι διεθνείς ελπίδες, κάτι που οδήγησε σε περισσότερη απογοήτευση ε, μπροστά σε για το ενδεχόμενο κατάρρευση και των δύο κρατών και την δυναμία της ε, διεθνούς κοινότητας να παρέμβει. Για να, το αποφύγουμε, για να αποφύγουμε περισσότερα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους άλλους παράγοντες περιοχής όπως η Ρωσία θα πρέπει ε, ε, να ε, παρέμβουν. Ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και τις δύο χώρες για ένα, μια ισορροπημένη λύση, ε, την υιοθέτηση των βασικών αρχών και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και την ανθρωπιστική κρίση, δεδομένου ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένους πληθυσμούς, αυτοί θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο η μόνη λύση είναι ο διάλογος και ο συμβιβασμό ε, με αλλαγή της νοοτροπίας ε, προκειμένου όλοι να σκεφτούν τις ανάγκες των υπολείπων και τα δεινά των λαών τους. Ε, η ειρήνη έφτασε στα Βαλκάνια, ήρθε ώρα να φτάσει και στον Νότιο Κάφκασο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τοκές. Για 1,5 λεπτό ο λόγος στον κύριο Σόπφλιν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή Εκπρόσωπε. Όπως φαίνεται από τη συζήτηση αυτή, η διαμάχη στον Αναγκόρο Καταμπάχα έχει παγώσει ε, εδώ και πολύ καιρό, αλλά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ε, να ξεπαγώσει και να πυροδοτήσει μια πολύ σημαντική κρίση. Το τέλος ε, του πολέμου του, μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμένια το 1994 οδήγησε ένα εκατομμύριο ανθρώπου στην προσφυγιά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που περιέπλεξαν τα θέματα. Η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν. Όλε οι χώρε αυτέ έχουν συμφέροντα στην περιοχή και ίσω αναμειχθούν αν ξαναξεσπάσει η σύγκρουση και αναθερμανθεί στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Το Αζερβαϊτζάν έχει ενεργειακό πλούτο και μπορεί τα χρήματα από το πετρέλαιο να τα χρησιμοποιήσει για να αποκτήσει στρατιωτικό εξοπλισμό τέτοιο, τέτοια προετοιμασία κάνει και η Αρμενία. Η Ρωσία προσπάθησε δυστυχώς ατυχώς στο Καζάν τον προηγούμενο μήνα να προωθήσει διαπραγματεύσει. Δεν υπάρχει μεγάλη βούληση από τι εμπλεκόμενε πλευρά, αλλά δυστυχώ έκβαση μέχρι στιγμή είναι η ματέωση, το αίσθημα τη ματέωση που είναι πολύ κακό σύμβουλο, ιδιαίτερα όταν ένα του πληθυσμού μια χώρα βρίσκεται υπό επίσημη κατοχή. Ε, το Αζερβαϊτζάν είναι απογοητευμένο από την ε, αντίδραση του υπόλοιπου κόσμου και ιδιαίτερα από την πρόσφατη ε, απόφαση για την προσχώρηση στο κίνημα των αδεσμεύτων. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση δεν αποκλείεται να έχουμε κάποια θερμά επεισόδια. Θα πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να συνεχίσουμε τις διαμεσολαβήσεις και τις διαπραγματεύσεις και είμαι υπέρ της θέσης για την ενεργό ανάμειξη στην ειρηνευτική επίλυση για της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Σέπφλιν. Το λόγο έχει 1,5 λεπτό κύριο Σκέλαμ. Κυρία Άστον, πρώτα απ' όλα λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή η συζήτηση δεν κατέληξε σε ψήφισμα. Η κατάσταση σήμερα είναι απαράδεκτη και απαιτεί επιγόντως μια ειρηνική και διπλωματική λύση. Πρέπει λοιπόν να προειδοποιήσουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι ως έχουν τα πράγματα η χρήση βίας θα οδηγούσε σε απρόβλεπτες συνέπειες για το σύνολο της περιοχής. Σήμερα δική μας ευθύνη είναι να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Ρωσία, να τους συστήσουμε να απέχουν από και να αμπλύνουν την ένταση. Η ευθύνη της Ρωσίας είναι μεγάλη γιατί πουλάει όπλα και στα δύο μέρη και η Μόσχα μοιάζει να ενδιαφέρεται να μακροημερεύσει η σύγκρουση, η ένταση. Χαιρετίζω το γεγονό ότι είπατε εκπρόσωπο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα. Γιατί πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διδραματίσει σημαντικό ρόλο. Αυτό όμω που χρειαζόμαστε σήμερα είναι η δέσμευση Ευρωπαϊκή Ένωση σε ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Μέχρι πρόσφατα λοιπόν ε, δεν υπήρχαν κίνητρα για ειρήνη. Όμω ε, είναι απαραίτητο για την αξιοπιστία μα στην περιοχή όχι μόνο να δείχνουμε στράτε αλλά και υπευθυνότητα απέναντι σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Καταρχήν και πρώτα απ' όλα πρέπει να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής από την περιοχή. Για 1,5 λεπτό λόγο στον κύριο Μπάτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τον Οκτώβριο 2010 είχα την ευκαιρία να πάω στον Αγκόνο Καραμπάχ και να συναντήσω και τις αρχές και τους πρόσφυγες. Σήμερα όμως διαπιστώνω την κλιμάκωση της ε, βία στην περιοχή ε, και ε, ένα αγώνα εξοπλισμού το Μίνσκ μάλιστα έχει αρχίσει να παίζει πιο σημαντικό ρόλο και με τη σύνολο κορυφή του Καζάν ε, από την άλλη μεριά διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά για να βρούμε μια ε, λύση. Μάλιστα η ρητορική του κ. Αλίεφ ε, οξύνει την κατάσταση. Σας υπενθυμίζω ότι οι τρεις πρόεδροι της ομάδας του Μίνσκ υπέβαλαν στο G8 της Ντοβίλ ένα οδικό χάρτη με έξι βασικές αρχές για την ειρηνική επίλυση του, της σύγκρουσης πρέπει να περάσουμε πια στην εφαρμογή τους και χωρίς την ε, συμμετοχή και εκπροσώπων του Ναγκόνο Καραμπάχ θα είναι δύσκολο να βρούμε μια μόνιμη λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της θα πρέπει να παρέμβει με διπλωματικά μέσα μέσω της ομάδας του Μίνσκ αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίξει και, τον, και τους αμάχους με βοήθεια προς τους ε, πρόσφυγες όπως κάναμε και στην Αυχαζία το 2008 για να προστατεύσουμε τον τοπικό πληθυσμό. Ε, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Καλό και την Προνική Προεδρία ε, που καθόρισε ότι, που το, την εταιρική σχέση της Ανατολής ως βασική προτεραιότητα ότι θα πρέπει να λάβει και αυτή δράση. Ε, η... Ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, ψηφίσει ένα, θα υιοθετήσει ένα ψήφισμα πιο ισχυρό από αυτό του κ. Κυριλόφ. Ο λόγος για 1,5 λεπτό στην κυρία Βάιντερε. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πριν τις θερινές διακοπές θα ήθελα να εξασφαλιστεί ότι στον Αγκόρνο Καραμπάχ δεν θα δούμε επανάληψη της κατάστασης της γεωργίας όπως είχε συμβεί, δηλαδή αυτά που είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 2008. Όμως ε, η κατάσταση της ε, περιοχής είναι ανησυχητική. Είναι κρίμα λοιπόν που ε, δεν θα υιοθετηθεί ψήφισμα πλευρά του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αρκετά δραστήρια στην αναζήτηση της λύσης για αυτό αυτή τη σύγκρουση. Έχουμε τα μέσα και έχουμε και την εμπειρία. Κύριε Άστον, η παρουσία σας στην ε, περιοχή θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο ρόλος της Ρωσίας ε, βέβαια είναι πολύ σημαντικός γιατί παρέχει εξοπλισμό και ε, εκπαίδευση στο Αζερβαϊτζάν. Ε, μετά τη συνοκορυφή του Καζάν, ο πρόεδρος Μετβέντεφ πέγραψε μια συνθήκη η οποία θα παρατείνει τις στρατικές επιχειρήσεις ε, της Ρωσίας στην ε, περιοχή μέχρι το 2042. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι και άλλες χώρες έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Χρειάζεται λοιπόν μια διεθνής παρουσία και μια διεθνής δράση όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις, ε, τις χώρες της ομάδας του Μίνσκ. Ε, θα πρέπει η, ε, η κατοχή να σταματήσει και οι πρόσφυγες να έχουν την ευκαιρία να γυρίσουν στα σπίτια τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να, όλη αυτή η διαδικασία να παρακολουθεί από διεθνείς παρατηρητές και να προσφύγουμε στο δημοψήφισμα. Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λίσεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπατή, εκπρόσωπε, θα ήθελα να πω ότι από τους προλαλήσαντες άκουσα πολλές προσδοκίες, υψηλές προσδοκίες από την Πολωνική Προεδρία σε ό,τι αφορά την σύγκρουση αυτή. Αλλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τις προσπάθειες της ΥΠΑ εκπροσώπου, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας ε, εκχωρεί όλες τις αρμοδιότητες για την εξωτερική πολιτική στην ΥΠΑ εκπρόσωπο. Δεν ε, ευθύνεται τόσο η κάθε Προεδρία. Πάντω γνωρίζω και προσωπικά τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Σικόρσκι, και είμαι 100% βέβαιο ότι ο κύριο Σικόρσκι, ο Πολωνό Υπουργό Εξωτερικών, θα υποστηρίξει τι δραστηριότητε τη κυρία Άστον μα ανησυχεί η κατάσταση στον Αγκόνο Καραμπάχ, αλλά υπάρχουν κάποιες κοντινέ μας περιοχές που δεν δημιουργούν μόνο ανησυχίε, αλλά και φρίκη. Για παράδειγμα, είμαι ο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γεωργία και πρόσφατα μετέβη στη χώρα αυτή. Συναντήθηκα με πολιτικούς, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον ΙΠΕΞ, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και όλοι είπαν ότι βλέπουμε φρικαλαιότητα από αυτά που μπορεί να συμβούν στον Αγκόνο Καραμπάχ γιατί δεν θέλουν καν να φανταστούν, να διανοηθούν τι συνέπειες θα έχει για την γεωργία μια έκρηξη αυτού, αυτής της σύγκρουσης. Γι' αυτό θα ήθελα να θερμοπαρακαλέσω την επατεκπρόσωπο να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα αυτό, συνεχίζοντας διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν, την Αρμενία αλλά και τη Ρωσία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λίσσα και για 1,5 λεπτό τώρα το λόγο έχει η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέδη Άστον, θα ξεκινήσω λίγο παλιότερα από την συνάντηση του Καζάν, θυμίζοντας σας ότι αν η εξέγερση του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ γινόταν σήμερα, παράλληλα με τις εξεγέρσεις των αραβικών λαών εναντίον τυραννικών και άδικων καθεστώτων, είμαι σίγουρη πως θα είχε την αμέριστη συμπαράσταση μας και την ενεργό στήριξη της ευρωπαϊκής κοινότητας. Το ίδιο θα συνέβαινε και στο Ναχίτσεβάν, μια περιοχή με πανομοιότυπο αυτόχθονα πληθυσμό αν εξακολουθούσε να υφίσταται εκείνος ο πληθυσμός. Αλλά δυστυχώς έχει εξαφανιστεί. Ανταυτού εκείνο που παρακολουθούμε σήμερα, εκείνο που βλέπουμε σήμερα είναι μια επιδιδευμένη ουδετερότητα ε, για την κατάσταση και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αμέτωχη ενώ μας ενοχλεί μόνο η πηγή των εξοπλισμών. Και δεν λέω βαρώνει Άστον ότι πρέπει να στείλουμε βομβαρδιστικά στον Κάφκασο. Απέναντία πρέπει με κάθε τρόπο να στηρίξουμε ενεργά την ειρηνευτική διαδικασία με εμφανή και ουσιαστική παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Κάφκασο. Από την άλλη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθούμε το Αζερβαϊτζάν που καταγγέλθηκε πολλέ φορέ διεθνώ και ειδικά στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού για την Συνεργασία και την Ασφάλεια στην Ευρώπη να ακολουθεί μια τρομακτική εξοπλιστική προσπάθεια βλέπουμε την κυβέρνηση του αζερβαϊτζάν αντί να αγωνίζεται για την ανάπτυξη και την ευημερία του αζερικού λαού έχοντα στη διάθεση τη τεράστιο ορυκτό πλούτο να τον δαπανά για εξοπλισμού. Και από την άλλη μα ανησυχούμε βεβαίω, γιατί τώρα μπήκε στην κούρσα των εξοπλισμών και η Αρμενία, μια χώρα που τελεί υπό οικονομικό εμπάρκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υφίσταται ένα άγριο εμπάρκο από όλε τι γειτονικέ τη χώρε και βεβαίω η αρμενία οφείλει να αποχωρήσει από κατεχόμενα εδάφη από το παιδινό ε, καραμπάχ όπω οφείλει να αποχωρήσει και η κύπρο, αλλά νομίζω ότι όλα θα πρέπει να επιληθούν στη βάση του δικαίου και όχι στη βάση του από που αγοράζει ο καθένα του εξοπλισμού. του. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Θεοχάρου, Για 1,5 λεπτό το λόγο έχει η κυρία Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, εγώ εκπροσωπώ σήμερα τη Σουηδία, αλλά πρέπει να σας πω, εγώ είμαι πρόσφυγας από τη Βοσνία. Έζησα λοιπόν τον πόλεμο στη Βοσνία και αυτά που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι εδώ σήμερα. Ήμουνα λοιπόν στη Βοσνία και περίμενα κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Αμερική, από τον Άτομο μα κάποιος, έστω κάποιος, να επέμβει, να κάνει κάτι, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Αυτή λοιπόν η απογοήτευση που βίωσα τότε με οδήγησε στο να ασχοληθώ με την πολιτική. Και αυτό που βλέπω σήμερα στο Ναγκόρνο Καραμπάχα είναι ακριβώς ε, το ίδιο σενάριο, επαναλαμβάνεται, ε, εδάφη υποκατοχή, εκτοπίζονται πολίτες, ε, γίνονται πρόσφυγες, μετά στις περιοχές αυτές εκφράζεται το αίτημα της αυτοδιάθεσης. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Βρίσκομαι εδώ και απαιτώ οι άνθρωποι να μην ζουν πλέον υποκατοχή. Και μόνο εφόσον θα έχουν επανέλθει πρόσφυγες στις αιστείες τους, μόνο τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για τελεσίδικες λύσεις. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται δημοψήφισμα αφού έχουν ήδη εκτοπιστεί οι πρόσφυγες. Πρώτα να επανέλθουν οι πρόσφυγες και μετά να συζητήσουμε για την ουσία των Κόνο Γιατί αλλιώς θα ζήσουμε για άλλη μια φορά τη Ρεπούμπλικα Σπέρσκα και αυτό δεν το θέλουμε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο Κάτσι ή ε, μάλλον πριν το ΚΑΤΣΔΙ, ο κύριο Στογιανόφ σήκωσε μπλε κάρτα. Δέχεστε την ερώτηση, κύριε Μπρισάτζιτ. Φυσικά, φυσικά, βεβαίω. Κύριε Στογιανόφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπρισάτζιτ, αν θυμάμαι καλά, η χώρα σα αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου και το Κωσυφοπαίδιο ήταν ε, μια περιοχή που αποσπάστηκε από κυρίαρχο κράτο. και όμω το αναγνωρίσατε θεωρώντα ότι είναι απολύτω νομότυπο ενώ αυτό που συμβαίνει στον αγώνο Καραμπάχ ε, αποτελεί αντικείμενο συζήτηση. Θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά γιατί μιλούμε για εθνοκάθαρση. Τι γνώμη έχετε για την ε, εθνοκάθαρση που έκανε το Αζερβαϊτζάν εις βάρος της Αρμενίας με όλο τον πληθυσμό του Μπακού. Κύριε Μπρισάτζιτς. Θα πρέπει να γνωρίζει ο κύριος Στογιάνοφ, κύριε Πρόεδρε, ότι το κοσυφοπαίδιο είναι, είναι ένα διεθνώς αποδεκτό και εξαιρετικό παράδειγμα. Η διεθνή κοινότητα δέχτηκε ως εξαιρετική και έκθετη την κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο και δεν δημιουργείται δεδικασμένη προηγούμενο για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς στην προσέγγιση μας. Όταν μιλούμε για υπερδυνιστερία ή για οπουδήποτε αλλού, τασόμαστε υπέρ τη ε, εδαφική ακαιρεότητας, της Γεωργίας για παράδειγμα, της Μολδαβίας. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συνεπής ε, στη θέση της και να προστατεύσει και την εδαφική ακαιρεότητα του Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστούμε κύριε Μπισάτζη. Τώρα περνάμε στο γύρο του Κατσδιάη. Το λόγο έχει πρώτα ο κύριο Λαντσμπέργκη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπη, αγαπητοί συνάδελφοι. Φαίνεται ότι η διαδικασία ανάλυσης των παγωμένων συγκρούσεων στην Αρμενία και στο Αζερβαϊτζάν φτάνει και μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται ότι εθελοτυφλούσαμε μέσα τις τουρθοκαμίνους και κρυβόμαστε και με τα σχήρας μας μπροστά στην ομάδα του Μίνσκ. Είχαμε όμω έναν 20 διάλογο που δεν κατέληξε πουθενά. Τελικά είναι καλύτερο αυτό από, από τον πόλεμο. Η στρατιωτική χρήση όμως εξακολουθεί να συνεχίζεται. Ο καρκίνος του πολέμου ήδη υπάρχει στην περιοχή και συνεχίζει, επιδεινώνεται η νόσος γιατί υπάρχει, ε, υπάρχουν δολοφονίες από σνάιπερς των εχθρών. Ας μην γελιόμαστε λοιπόν. Ε, η ερώτησή μας είναι να δράσει κανείς ή να μην δράσει. Το θέμα δεν είναι πόλεμος ή όχι. Θα πρέπει να καλύψουμε και να είμαστε άτεκτοι, να καλύψουμε τη διαπραγμάτευση ε, να λάβουμε υπόψη το κατεχόμενο έδαφος του Αζερβαϊτζάν, τους εκτοπιστέντους, τους πρόσφυγες, στην, τα προβλήματα επικοινωνίας του Αζερβαϊτζάν. Θα πρέπει να αντιληφθούμε πλήρως την κατάσταση και να έχουμε σοβαρές συζητήσεις με τη Ρωσία για το ρόλο που έπαιξε στην περιοχή. Ευχαριστούμε κύριε Λασμπέργης. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Νίτρας. Ευχαριστώ. Ε, ο Νότιος Κάφκασος είναι μια περιοχή που σε κάθε γωνιά του δρόμου βλέπουμε πρόσφυγες. Από το Αζερμπαϊτζάν, από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, από την Γεωργία, την Απχαζία, την Νότια Οσετία. Αλλά ακόμη και στην Αρμενία είδα πρόσφυγες. Όχι από τον Αγκόρνο Καραμπάχ, από τον Μπακού έχουν και κάποιο δρόμο δικό τους ε, που το λένε Μπακού. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι αν ε, ε, δείξουμε μεροληψία σε αυτή την σύγκρουση, αν ταχθούμε με το πλευρό του ενός μόνο, δεν μπορούμε να μιλούμε για θετική δράση στην περιοχή αυτή. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι όλες αυτές οι συγκρούσεις έχουν ένα κοινό παρανομαστή, τον σοβιετικό υπεριαλισμό. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Εγώ δεν πιστεύω στα σχέδια της ομάδας Μίνσκ και στην πρακτική συμβολή της με αυτή τη μορφή. Η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει στην διευθέτηση τη σύγκρουση αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο πραγματεύση με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία, ε, ε, ο ρόλο τη θα ενισχυθεί περισσότερο. Κυρία ε, είπατε εκπρόσωποι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα πρέπει να το αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα στα καθήκοντά σας τον επόμενο καιρό. Ευχαριστώ για ένα λεπτό το λόγο κύριο Στάνοκ. Το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ ε, χαρακτηρίζεται παγωμένη σύγκρουση πολύ συχνά, αλλά λιώνει πολύ γρήγορα ε, με τους ελεύθερους σκοπευτές ε, και διάφορα άλλα επεισόδια τα οποία κλιμακώνουν την κατάσταση, αυξάνουν τα θύματα και υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει πόλεμος με το Ιράν, τη Ρωσία από την μία μεριά και, τη Ρωσία, και την Τουρκία από την άλλη. Και βέβαια πολλά τεράστιο αριθμό πετροδολαρίων ε, χρηματοδοτεί αγορά ε, εξοπλισμού και ε, την κόρσα των εξοπλισμών κάτι που οδηγεί το Αζερβαϊτζάν να αυξήσει την ισχύ του αντί της μικρής Αρμενίας και να προσπαθήσει ενδεχομένως να πάρει πίσω τον Αγκόνο Καραμπάχ. Η Αρμενία σίγουρα θα πρέπει να αποσυρθεί από τη γύρω περιοχή του, Ναμπόρν, του Ναγκόρνο Καραμπάχ και να επιτρέψει στους προφύγες να επιστρέψουν στα ε, σπίτια τους. Ε, ούτε η αυτοδιάθεση, ούτε η εδαφική κυριαρχία είναι απόλυτες αρχές. Όλοι θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι στην εξωτερική πολιτική. Συνεπώς, ε, ε, κάνω έκκληση μετά την αποτυχία του Καζάν στα μέρη, στα ενδιαφέρομενα μέρη, να προσπαθήσουν μεταξύ του να λύσουν τα πρόβλημά τους με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, και λέω σε εσάς κύριε Άστον, ε, είναι ευκαιρία σας να κερδίσετε ένα, το βραβείο Νομπέλ της Ειρήνης. Για ένα λεπτό ο λόγος στην κυρία Μπασέσκου. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Declarația înaltului reprezentant completează inițierea reformei. Η ανακοίνωση της ΕΠΑ της εκπροσώπου συμπίπτει με την ανθεώρηση της ανατολικής πτυχής της, εταιρικής, της σχέσης γειτονίας. Ε, και τον Αγώνο Καραμπάχ και η Περνιστερία αποτελούν ε, προτεραιότητες ε, προκειμένου να εξασφαλίσουν σταθερότητα στα εξωτερικά μας σύνορα. Παρόλη την ανακοχή που υπογράφηκε το 1994, οι εντάσεις κλιμακώνονται οι διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα με την υποστήριξη ομάδα του Μίνσκ έφτασαν σε ένα κρίσιμο στάδιο. Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής του Καζάν ε, δεν βελτίωσε τις σχέσεις ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία. Αντιθέτως, η αντίδραση ήταν μια κούρσα των εξοπλισμών ε, και η πόλωση ε, Ελπίζω ότι η ομάδα του Μίνσκ θα βρει μια λύση αποδεκτή και από, τα δύο, και τις δύο πλευρές ε, γιατί οι ε, ε, νέες εχθροπραξίες θα μπορούσαν να, υποσκάψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενεργειακή της ε, επάρκεια. Κύριος Μπέλτερ, για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω θα έπρεπε να παίξει πιο ενεργό ρόλο στον Αγκόρνο Καραμπάχ Μακάρι η Λέιδη Άστο να πάρει το βραβείο Νόμπελ αν να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ε, το... Ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν όμως, θα μπορούσατε να με ενημερώσετε. Γιατί μετά την αποτυχία των συνομιλίων του Καζάν, της συνομιλίας του Καζάν, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είπε ότι αυτό αυτή η περιφερειακή σύγκρουση θα πρέπει να λυθεί από τους ενδιαφερόμενους της ίδιας περιοχής, τα μέρη της ίδιας περιοχής. Ο λόγος για ένα λεπτό στην κυρία Βαϊντέρε. Ε, I'm very sorry. I just wanted to make... Ε, λυπάμαι πολύ. Ήθελα να κάνω μια διόρθωση γιατί οι συνάδελφοι που άκουσαν την ομιλία μου στα αγγλικά μου επισήμαναν ότι κάτι που είπα ίσως ε, να μην ερμηνεύτηκε σωστά. Θέλω να επαναλάβω λοιπόν κάτι. Η Ρωσία δίδει στην Αρμενία όπλα και ε, στρατιωτικό εξοπλισμό και όλα τα άλλα υποθέτω ότι μεταφράστηκαν σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, διευκρίνηση. Η κυρία Άστον έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι ε, ιδιαίτερα σύντομη γιατί νομίζω ότι τα σημαντικότερα ελέγχθησαν στις ε, παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ και εγώ πράγματι ε, έχει φτάσει στιγμή να μεταβώ στην περιοχή. Ίσως έπρεπε ήδη να έχω πάει αλλά υπήρχαν τόσα γεγονότα και για μένα είναι μια προτεραιότητα αυτή να μεταβώ στην περιοχή για να διασφαλίσω ότι εκπέμπουμε το σωστό μήνυμα. Θέλω να έχω συζητήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και των δύο χωρών ε, και με τους επικεφαλείς της ομάδας του Μίνσκ. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι θα χαρώ πάρα πολύ το να μπορέσω να παίξω σημαντικότερο ρόλο. Η Γαλλία επιθυμεί διακαώς να συνεχίσει το ρόλο που παίζει, πιστεύει ότι έχει να προσφέρει ακόμα πάρα πολλά. Ο δικός μας ρόλος είναι να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη και να προσφέρουμε ε, και την ε, σωστή υποστήριξη. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν από τους αξιότιμους βουλευτές ότι πρέπει κανείς να ασχολείται όχι μόνο με τα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και με την καθημερινότητα, με τα καθημερινά ε, προβλήματα. Να υπάρχει η ανθρώπινη επαφή. Όπως είπαν και οι αξιότιμοι βουλευτές δεν είναι παγωμένοι αυτή η σύγκρουση ε, αρχίζει πάλι να θερμαίνεται και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Ε, ανησυχώ με αυτό που ότι είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο της εμπιστοσύνης. Ε, θεωρώ ότι η συζήτηση λαμβάνει η χώρα την κατάλληλη στιγμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό γιατί είναι ένα θέμα που το γνωρίζουμε πολύ καλά στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να συνεργαστούμε με όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην ομάδα Μίνσκα και ο λόγος που θέλουμε να στείλουμε ένα νέο απεσταλμένο είναι γιατί θέλουμε να καταβάλουμε μεγαλύτερε ε, προσπάθειες, βεβαίως παράλληλα και με όλα τα άλλα θέματα που τρέχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με μεγάλη μου χαρά θα παρακολουθήσω τη συνέχιση της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε κυρία Άστον. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη δήλωση της ΥΠΑΣ εκπροσώπου για εξωτερικά θέματα και κοινή εξωτερική πολιτική με θέμα τις προπαρασκευαστικές δράσεις για τις βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία, για τη, Ρωσία, για τη...